ενθεί στη νομική επιτροπή που είναι αρμόδια καθήλια για τα θέματα αυτά. Επίσης, η αρμόδια καθήλια επιτροπή ε, μου έθεσε ένα ερώτημα για ψήφισμα δεύτερης ανάγνωσης που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινή συνόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού θα θεωρηθούν εγκεκριμένες αυτές οι διατάξεις αν ε, στην ε, γνωστή προθεσμία δεν υποβληθούν ε, προτάσεις για την διεξαγωγή ψηφοφορίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στα σοβαρά θέματα, δηλαδή στην διάταξη των εργασιών που έγινε δεκτή από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων ε, στη συνεδρίαση της 5ης 10ης ε, Σεπτεμβρίου με βάση το σχετικό άρθρο του κανονισμού και έχετε λάβει αυτή την ε, διάταξη των εργασιών, το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Βλέπετε ότι το πρόγραμμα μας ε, είναι πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ακροάσει ε, των Επιτρόπων και θα ψηφίσουμε σήμερα για τις ε, εγκρίσει αυτών των διορισμών. Επίση, αύριο θα ακούσουμε την ομιλία για τις πολιτικές και τεχνικές προτάσεις ε, για την επόμενη κοινοβουλευτική, για την επόμενη θητεία του Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, έχουμε τις προτάσεις ε, του, της Σουηδικής Προεδρίας και σήμερα και την Τετάρτη θα μιλήσουμε και για τις αντιπροσωπείες. Το Συμβούλιο θα μας προτείνει και τον κανονισμό για το 2000, τον προϋπολογισμό για το 2010. Βλέπετε ότι η διάταξη των εργασιών μας είναι υπερφορτωμένη, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα τα θέματα με τη σειρά, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα έρθω στο σχέδιο μέρησης διάταξης. Απλώς έκανα κάποιες παρατηρήσεις. Και για κάθε σημείο μπορώ να σας δίνω το λόγο. Καταρχήν, για